Καλησπέρα σας. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία πρώτα της έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας του κυρίου Μέλλο με θέμα τον τομέα των απειροκυπευτικών ε, από τη μεταρρύθμιση του 2007 σήμερα. Παρακαλώ, εισηγητής, αν θέλει το λόγο μπορεί να τον πάρει. Κύριε Μέλο. Πρόεδρε, έχω μια, ένα αίτημα για, την, για το κατάλογο ψηφοφοριών. 123 τροπολογία λέγεται στον κατάλογο ότι είναι ανεξάρτητη από την 91. Εγώ θεωρώ ότι 123 Μάλλον λέγεται στον κατάλογο ότι εξαρτάται από την ψηφοφορία της 91. Ε, εγώ, συμφωνώ, εγώ θεωρώ ότι είναι ανεξάρτητη η ψηφοφορία της μιας από την άλλη. Η γραμματεία μου απήντησε ότι ε, έχει διορθωθεί αυτό στον, ε, θα έπρεπε να έχει διορθωθεί στον κατάλογο, οπότε αν θέλετε να την ψηφίσουμε ξεχωριστά την τροπολογία. 123 Πρόεδρε. Η γραμματεία Κύριε Τσούλο, επιβεβαιώνει το σχολείο σας. Έχετε δίκιο. Τώρα ο εισηγητής ο κύριος Μέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ασχέτως των αποτελεσμάτων και το ότι θα γίνει τελικός με αυτή την ψηφοφορία, ήθελα απλώς να παρατηρήσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είχαμε μια σημαντική μερίμνα για αυτή την έκθεση, να υπάρχουμε μέτρα καταπολέμησης των αθέμητων ε, πρακτικών που ζημιώνουν τους παραγωγούς και τους γεωργούς. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στη δεύτερη παράγραφο μία πολύ συγκεκριμένη μνήα και επίσης την τροπολογία 90 που οδεύει στην ίδια κατεύθυνση. Και εδώ οι τροπολογίες 84, 88 και 92 θα μπορούσαν να συνδυάσουν ε, κάποιες από τις ιδέες και της κυρίας ε, Μαγκίνες που αναφέρεται σε unfair trade practices. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο εδάφιο της ε, τροπολογίας 90 και επίσης να πω ότι το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές πρόεδρε επέβαλαν μια εναλλακτική τροπολογία στην τροπολογία 8 και οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές μαζί με τους φιλελεύθερους το ίδιο για την τροπολογία 9 μετά από συζήτηση με τους ε, σκιώδεις εισηγητές να πω ότι θα αποσύρουμε την 8η τροπολογία δεχόμενη την ένατη των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών διότι είναι πολύ σημαντικό να ε, είναι ισχυρή έκθεση και να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή συνένεση ώστε να αποσταλούμε και ένα θετικό ε, μήνυμα προς την Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Περνάμε στην ψηφοφορία. Όταν έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία θα σας ενημερώνω εγκαίρως. Τροπολογία 78. Ψηφίζουμε διανατάσεις της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 80. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 79. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 77. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 82. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται η προηγούμενη. Εγκρίνεται. Κατά. Εγκρίνεται. 83. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 85. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Αυτό είχα πει. Τροπολογία 88. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ίδιο αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 86. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτή απορρίπτεται. 87. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 89. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. αν διαπιστώνω ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι υπέρ, δεν πρόκειται να ρωτώ καν αν κάποιο είναι κατά. Θεωρώ ότι εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Ποιο είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 92. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά. Τροπολογία 93. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 94. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 97. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 97. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 95. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 96. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 98. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Έχω την αίσθηση ότι εγκρίνεται, αλλά ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται τελικά. Συμβαστική τροπολογία 6. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Κατάλληλο, πρόεδρο. πρόεδρος. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 103. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ. Σηκώστε τα χέρια παρακαλώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της πέμπτης τροπολογίας της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ της ε, τροπολογίας 8 τη Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. Δύσκολο να το δει κανείς με τα χέρια. 104. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 105. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 106. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 107. Ποιος είναι υπέρ. 107 και όχι 115 που είπε ο πρόεδρος. 107 λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 115. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 112. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 110. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 111. Υπέρ. Εγκρίνεται. 108. Υπέρ. 113. Μπούντα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 117. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 116. Ποιος είναι υπέρ. Εκατόν δεκαοκτώ λέει γραμματεία τώρα. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο, πρέπει να πάμε κατευθείαν στην 118. Ποιο είναι υπέρ τη 118. Κατά. Εγκρίνεται. 114. δεκατέσσερα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 119. δεκαεννέα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 120 υπέρ. Εγκρίνεται. Εκατόν είκοσι ένα υπέρ. Εγκρίνεται. Εκατόν είκοσι δύο. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 122. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 123. Ποιος είναι υπέρ? Ποιος είναι υπέρ της 123. Κατά. Απορρίπτεται. 124. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 125 υπέρ. Εγκρίνεται. 126. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 127. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού υπέρ. Εγκρίνεται. 129. Ποιος είναι υπέρ. Μα αυτό είπα λέει ο πρόεδρος. 129. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 130. Ποιο είναι υπέρ της τροπολογίας 130. Εγκρίνεται και αυτή. 131. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 84. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 84. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 132. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 133. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 134. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 135. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ της κοντ. Κατά. Απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε για καλό και για κακό. Τροπολογία 7 της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ε, εγκρίνεται με τέσσερι ψήφου διαφορά, αλλά καλά που το ελέγξαμε. Επόμενη 126, 136 ποιο είναι υπέρ, εγκρίνεται. 137 ποιο είναι υπέρ, εγκρίνεται. Κοντ 9 ποιο είναι υπέρ. Κατά. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 9 της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 140. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 139. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 142. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 142. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 144. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 100 138. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 145. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 146. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 143. Ποιος είναι υπέρ. Ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 της κοντ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 147. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 148. Υπέρ. Κατά. Οριακή διαφορά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 148. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 149. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 149. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με την ίδια διαφορά. Τέσσερις ψήφους διαφορά μάλλον. Ποιος είναι υπέρ της 150. Κατά. Απορρίπτεται 151 υπέρ. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Εγκρίνεται. 154 υπέρ. Εγκρίνεται. 155 υπέρ. Εγκρίνεται. 156 υπέρ. Εγκρίνεται. 158 του κύριου Ταραμπέλα υπέρ εγκρίνεται. 159 ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 160 ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 161 υπέρ, εγκρίνεται. 168 ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 165 υπέρ, κατά Απορρίπτεται. 171 υπέρ. Εγκρίνεται. 164 υπέρ. Ή μάλλον 170. 70 λέει ο Πρόεδρος. Ποιος είναι υπέρ της 170. Εγκρίνεται. 163. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 162. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 172. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 169. 173, ναι, συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 174. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται, αλλά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 174. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 175. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 176. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 180. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 179. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 177. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 181. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 182. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 183. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 184. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 185. Ποιος είναι υπέρ? 187. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 189. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 186. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 188. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 190. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Ηλεκτρονική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τις συμβαστικές τροπολογίες θα τις ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 193. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 197. Ποιος είναι υπέρ της 197. Κατά. Απορρίπτεται. 198 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα της 198. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 200. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Α, όχι, πίπτη, συγγνώμη. Πάμε στη 204. Ποιος είναι υπέρ? 201. Η 204 εγκρίνεται. 201 επίσης εγκρίνεται. Τροπολογία 203. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 202. Ποιος είναι υπέρ. Όχι, όχι 202 καταπίπτει. Διακόσια πέντε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 205. Παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Ψηφίσαμε τη 205. Εγκρίνεται. 206. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 207. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 208. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 209. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 210 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 211 υπέρ. Εγκρίνεται. 212 υπέρ. Εγκρίνεται. Κοντ 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Κοντ 11. Αν θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 10 της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Κοντ 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Κοντ 12. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Κοντ 13. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Κοντ 14 λέει ο πρόεδρος. Ω, συγγνώμη. 16. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 2.13 του κυρίου Καπούτο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 213. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 219. Ποιος είναι υπέρ. 219. Κατά. Απορρίπτεται. 218. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 214. Ποιος είναι η... ή μάλλον... Πάμε στη 220. Ποιος είναι υπέρ. 2.20. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 221. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 2.22. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 1. Um... Πρέπει να ψηφίσουμε την 214 που την ξεχάσαμε. Ποιος είναι υπέρ? Όχι 14, 216. 214 έχει καταπέσει, μια και εγκρίναμε την 218. Αυτή που έμεινε να ψηφίσουμε είναι 216 και όχι 214. Δίκιο έχετε, δίκιο έχετε. Ευχαριστούμε. Ψηφίζουμε για την 216. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. ...216, συγγνώμη, πριν ήταν η 211, τώρα η 216. Μια στιγμή να το ξεκαθαρίσει η γραμματεία. Poprawka 217. 217 λέει ο πρόεδρος τώρα. Α, την ψηφίσαμε. 220. 220. Κατά. Απορρίπτεται. Γιατί δεν ψηφίζουμε τη 217, γιατί δεν την ψηφίσαμε. Η 219 κατα... καταψηφίστηκε, οπότε οφείλουμε να ψηφίσουμε τη 217. Α, το επιβεβαιώνει και η γραμματεία. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 217. Ποιος είναι υπέρ της 217. Κατά. Εγκρίνεται η 217. Τώρα, 200... Ποπράφκα νούμερα 1. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ποπράφκα numer 2. Παραμπούντι. Κτο είναι Κατά της, α, της α εγκρίνεται. Κοντ α, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, καταπίπτει. Τροπολογία 5, 5, ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 5, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία Β της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Ποιος είναι υπέρ. Κοντ Β. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 10. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. 24 προς 19 εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία τσέκεντε της κοντ. Ποιος είναι υπέρ των δύο τροπολογιών. Σίκεντι. Κατά. καταπίπτει, μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για τις τροπολογίες C και D της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Κοντ ε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Κοντ 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 3 της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Ποιο είναι υπέρ. 19, συγγνώμη. ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχο για την 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 23. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 30 το του κυρίου Ντεκάστρο. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Εγκρίνεται. 34 ή μάλλον όχι. Πάμε στην 36. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 40. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού ή μάλλον καταπίπτει αυτή. Πάμε στην 41. Προφορική τροπολογία του κυρίου Ταραμπέλα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Ακαταπίπτει, συγγνώμη. Πάμε στη 45. Ταραμπέλα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 53. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 54. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εξήντα ένα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Εξήντα δύο. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 64 υπέρ, εγκρίνεται. 63 υπέρ, ή μάλλον καταπίπτει 63. 65, 67, ποιος είναι υπέρ, υπέρ της 67, εγκρίνεται. 68, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 70, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 69. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 71. Υπέρ. Κατά. Απο, ε, απορρίπτεται. 72. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 72. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 73. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 74. Υπέρ. Εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 76. Υπέρ. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος όπως έχει τροποποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Χωρίς ψήφους κατά, συγχαρητήρια κύριε Νονομέλο, εγκρίθηκε η έκθεσή σας. Ο εισηγητής. Πρόεδρε, πολύ σύντομα να πω ότι είναι θαυμάζια τα αποτελέσματα και να ευχαριστήσω όσου εργάστηκαν σκληρά για να είναι έτοιμε οι και όσου συμμετείχαν στι διαπραγματεύσει. Κυρίως να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας από την γραμματεία του ΕΛΚ, ε, τους σκιώδεις εισηγητές διότι ήταν εργατικοί και είχαν συμφιλωτική διάθεση στην όλη διαδικασία. Και νομίζω ότι πλέον με, την, τα μέτρα αυτά θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στις οργανώσεις παραγωγών κάτι χρήσιμο ε, και από την πλευρά του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και επιτέλους θα δείξουμε την διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευκολύνει τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε θερμά και θερμά συγχαρητήρια και σε εσά και στους συνεργάτες σας και σε όσους σας βοήθησαν. Τους συμβούλους, βοηθούς, γραμματεία κλπ. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. που αφορά την κατεξοδότηση, τον κατεξοδότηση κανονισμό για το αλκοόλ. Ε, με βάση το άρθρο 105 του κανονισμού ε, έχουμε καταξιδότηση πράξη μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, 20 Φεβρουαρίου. Και προβλέπεται με βάση το 105.3 την ε, χρήση εθνικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και αντικαθιστά, καταργεί μάλλον τον κανονισμό 200, 2336 2003 για καθορισμό ορισμένων λεπτομεριών της εφαρμογής ε, του κανονισμού 670 του 2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της εθιλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης. Ψηφίζουμε το προήμιο πρώτα. τα επιμέρους στοιχεία του προημείου θα ψηφίσουμε. Το το Ποιος είναι υπέρ του σημείου α στο προημείο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτω. Σημείο β. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Σε, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Δελ, D, E και F μαζί, D, E, F μαζί, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνονται... Οπότε ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος, την πρόταση ψηφίσματος που απορρίπτει την κατεξοδότηση πράξη. Με ονομαστική κλίση θα ψηφίσουμε το, την πρόταση ψηφίσματος που απορρίπτει την κατεξοδότηση πράξη. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το ψήφισμα, οπότε απορρίπτεται η κατεξουσιοδότηση πράξη. Περνάμε στην ψηφοφορία της σύστασης ε, για τον κατεξοδότηση κανονισμό του ε, Απριλίου με βάση τον κανονισμο 13.05.2003 του κανονισμού, κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με θέμα τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική ανάπτυξη. Η Επιτροπή ζήτησε να ψηφίσουμε την κατεξοδότηση αυτή πράξη προκειμένου να εγκρίνει τα προγράμματα ανάπτυξη πέθρου που περιμένουν στα κράτη-μέλη την έγκριση. Ψηφίζουμε υπέρ της κατεξοδότησης πράξης. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ. Μία ψηφοφορία κατέτσι του εισηγητού αναβλήθηκε. Η γνωμοδότηση για τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρήπων αναβλήθηκε μετά από αίτημα του εισηγητού του κύριου Χόιτεμα. Θέλετε να πείτε κάτι από αυτού, κύριου Χόιτεμα. παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, να σας πω απλώς ότι ακόμα διαπραγματευόμαστε με τους χιλιόδες και χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο για να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Είναι καλό να έχουμε λοιπόν μια στεναρή θέση ως άγκρη, οπότε θα χρειαστούμε και άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας ε, ενημερώσω και να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους του κυρίου Λίντς. Δυστυχώς γίνατε μάρτυρες ψηφοφορίας και όχι συζήτησης που είναι συνήθως πιο ενδιαφέρουσα, αλλά σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Περνάμε στο σημείο 14, το εμπόριο προϊόντων φώκιας. Συντάκτη γνωμοδότη είναι ο κύριος Βοητσεχόφσκι και αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή είναι η Επιτροπή Εσωτερική Αγορά και προστασία του Καταναλωτή. Εμεί θα συντάξουμε γνωμοδότηση. Δεν θα δώσω εγώ τις εξηγήσει. Ε, καλύτερα να το κάνει ο κύριος Κούσμιου, που είναι αντικαταστάτης του συντάκτη και γραμματότης του κυρίου Βουτσεχόφσκι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Βουτσεχόφσκι για την απουσία του αλλά έχει σημαντικές ανηλυμένες υποχρεώσεις ε, στην πατρίδα του και ε, μου, μου ανέθεσε να παρουσιάσω εγώ τη θέση του. Ο περιορισμός του εμπορίου προϊόντων φώκες ζητήθηκε εδώ και πολύ καιρό από, ε, από πολυάριθμες οργανώσεις για την προστασία των ζώων καθώ και από την κοινή γνώμη που δεν δέχεται να σφαγιάζονται, να θανατώνονται οι φώκες με απάνθρωπο και βιοτρόπο για εμπορικού σκοπού. Σύμφωνα με διάφορε επιστημονικέ έρευνε, οι φώκε είναι ζώα ιδιαίτερα ευφυή και ευαίσθητα, γεγονό που δικαιολογεί ακόμη περισσότερο την ανάγκη προστασία του έναντι τη σκληρότητα και τη ταλαιπωρία. Παράλληλα, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι τα προϊόντα φώκια δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ ε, δεν τα έχουν μεγάλη ανάγκη, μπορούν κάλλιστα να ζήσουν και χωρί αυτά. Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάζουσα κατάσταση των ε, Εσκιμών, των Ινουιτών και άλλων αυτόχθονων κοινοτήτων, για τους οποίους το κυνήγι της Φώκιας συνιστά μακροχρόνια παράδοση. Και είναι πολύ σημαντικές εισαγωγέ προϊόντων Φώκιας που θα πρέπει να περιοριστούν στα προϊόντα που προέρχονται από το κυνήγι στο οποίο επιδίδονται οι κοινότητε αυτέ. Ενώ παράλληλα θα πρέπει να απαιτούμε να τηρούν στο μέτρο του δυνατού τι υψηλότερε δυνατέ ανθρωπιστικέ προδιαγραφέ. Στην περίπτωση τήρηση αυτών, η Επιτροπή θα πρέπει να προσφύγει σε άλλα μη νομοθετικά μέτρα, προκειμένου να ευνοήσει τη διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά. Το θέμα του κατάλληλου ελέγχου τη τήρηση των ορίων που εφαρμόζονται στι αγωγέ προϊόντων φώκε αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο Δεδομένου ότι ο έλεγχο αυτό δεν θα είναι αποτελεσματικό παρά μόνο αν εισαγωγή των σχετικών προϊόντων υποχρεούνται να αποδείξουν ότι τα εν λόγω προϊόντα προέρχονται από τι κυνηγετικέ δραστηριότητε των ε, παραπάνω κοινοτήτων. Μέσω τη θέσπιση παρόμοιων απαιτήσεων, ο νομοθέτη υιοθετεί μια προσέγγιση που συμβάζεται με του βασικού βασικούς στόχου του κανονισμού, οι οποίοι υπακούν σε ηθικά κριτήρια σε ό,τι αφορά το κυνήγι τη φώκια για εμπορικού σκοπού. Ο εισηγητή κρίνει ότι θα πρέπει να προβρεθεί δυνατότητα προσωρινή θέσπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιας πλήρους απαγόρευσης εισαγωγή προϊόντων φώκες προερχόμενων από τρίτε χώρε, στι οποίε η θύρα πραγματοποιείται έκδηλα κατά παράβαση των προτύπων που απαιτούνται για τη μείωση του πόνου, τη αγωνία, του φόβου και άλλων μορφών ταλαιπωρία των ζώων που αποτελούν αντικείμενα του κυνηγιού αυτού. Σας ευχαριστώ. Αυτή ήταν η θέση του εισηγητού, του συντάκτου της γνωμοδότησης. Σας ευχαριστούμε κύριε Ευρωβουλευτά. Το λόγο ζήτησε πρώτα ο κύριος Ρόντε. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, τον συνάδελφο για την ε, παρουσίαση της θέσης του εισηγητού. Δεν είμαι σίγουρος αν ο εισηγητής έχει μείνει σταθερό στην ε, ε, ε, νομοθεσία που είχε ψηφιστεί από το 2009, αν βασίστηκε στην πρόταση της Κομισιόν και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την, το κυνήγι φώκιας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι παραδόσεις τηρούνται χιλιάδες χρόνια και τα προϊόντα ε, του δέρματος φώκιας ε, χρησιμοποιούνται εδώ και εκατοντάδες ε, χρόνια. Το κρέας της φώκιας καταναλώνεται. Η φώκια συνδέεται με μεγάλη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την οικονομία των Ινουητών. Εμείς τι κάνουμε, είμαστε εντελώς αντίθετοι σε όλα όσα μπορούν να βοηθήσουν ίσως κάποιες μειονοτικές ομάδες. Ήδη από το 2009 είχαμε την, το, την απαγόρευση των, της χρήσης τέτοιων προϊόντων και αυτό είχε πολύ σημαντική επίπτωση στις, στην κοινωνία των εννοητών. Φυσικά είναι μια εξαίρεση αυτό. Αλλά βεβαίως δεν έχει μειωθεί και δεν έχει μειωθεί ε, έχει μειωθεί μάλλον ο αριθμό των κυνηγών στη Γρυλανδία εδώ και περίπου ένα, ε, κατά ένα τρίτο και πλέον το εισόδημά του είναι ένα τρίτο μικρότερο, χαμηλότερο από ό,τι ήταν παλιά. Αυτό σημαίνει ότι οι Ινουίτες έχουν μειώσει και το κυνήγι κατά 50%. Παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς εμπειρογνώμονες λένε ότι θα μπορούσαν οι Ινουίτες να ε, κυνηγήσουν τρεις φορές περισσότερες ε, φώκες και παρόλα αυτά να υπάρχει βιώσιμο κυνήγι φώκιας. Και η, και η Greenpeace το λέει ότι το κυνήγι φώκιας είναι βιώσιμο. Επίσης, ε, η Γενική Γραμματεία του WWF λέει ότι το κυνήγι φώκιας είναι βιώσιμο και ότι η φώκια είναι ένα ζώο αρκετά αγαπητό, κάνει τον κόσμο να χαμογελάει, ζει σε ένα πολύ μοναδικό βιότοπο και φαίνεται πως είναι πολύ ευαίσθητο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα ζώο που είναι πολύ αγαπητό στον κόσμο. Και το αποτέλεσμα της έκθεσης είναι ότι το κυνήγι της ε, φώκιας είναι βιώσιμο. Η Κομισιόν τώρα έρχεται και αφήνει όλη την επιστημονική έρευνα, όλη την ιστορία, όλους τους, όλες τις παραδόσεις, τα παραγωνίζει όλα αυτά και ξέρω ότι και ένας Σουηδός υπουργό που ήταν πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, επιτέθηκε στους ε, Ινουίτες που ε, κυνηγούν φώκε. Εγώ ω Δανό είμαι πραγματικά αντίθετο με το απαγόρευση που έχει τεθεί από το 2009. Οι φιλελεύθεροι έχουν θέσει το θέμα αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε σε διέξοδο και δεν βλέπω και φως στο τούνελ. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις από τον ΠΟΕ για, το, για την απαγόρευση του κυνηγιού η απαγόρευση δεν θα έρθει του 2009, η Κομισιόν όμως πρέπει παρόλα αυτά να αντιδράσει. Ήδη έχουν αρθεί κάποιες αρκετά σημαντικές εξαιρέσεις και ήδη έχουν μπει στην, στα κείμενα αυτά και κάποια σημεία που στιγματίζουν την κοινότητα των, των Ινουητών. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει, έτσι ώστε να συνάδει με τις πρακτικέ στην περιοχή. Όλοι βεβαίω είναι υπέρ τη καλύτερη ενημέρωση για το κυνήγι τη φώκιας. Και είμαστε αντίθετοι του να μην αρθούν οι ε, εξαιρέσεις ή οι ε, ρήτρε αναθεώρηση. Αυτές οι αποφάσεις ήταν ε, νομίζω αρκετά αυθαίρετες στον τρόπο με τον οποίο πάρθηκαν. Είναι απογορευμένο βεβαίως να σκοτώνει κανείς ε, ε, φώκες μικρής ηλικίας. Δεν μιλούμε για αυτό φυσικά. Αλλά μιλούμε για κάποιες κοινότητες οι οποίες έχουν επιβιώσει ακριβώς πάνω σε αυτό. Οι κυνηγοί φώκες δεν μπορούν να ε, αλλάξουν ξαφνικά επάγγελμα και να βρούνε μια άλλη δουλειά. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χάζεκαμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή που έχει συντάξει μια πολύ σαφή έκθεση αλλά ας είμαστε Το κόμμα για την υπεράσπιση των ζώων που εκπροσωπώ δεν κάνει καμία διάκριση για την παραγωγή ουδήποτε προϊόντος από ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι γούνα είτε οτιδήποτε άλλο ε, και από φώκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς όμως ο ΠΟΕ που ε, λαμβάνει υπόψη μόνο κοντόφθαλμα εμπορικά συμφέροντα, τη στιγμή αυτή και παρά την απαγόρευση προϊόντων ε, που παράγονται από τα ζώα αυτά, προβλέπει δύο εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις για τις ε, και τις αυτόχθονες κοινότητες, κοινότητες αυτοχθόνων, που δεν έχουν εμπορικές σχέσεις μόνο μαζί μας προφανώς. Εμπορεύονται και με άλλους εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτή η εμπορική, αυτός ο εμπορικός όγκος μπορεί να είναι σημαντικότερος από ό,τι φανταζόμαστε. Παρόλο που στην Ευρώπη υπάρχει απαγόρευση εμπορίας ε, δερμάτινων από φόκια, και γούνα φώκιας για λόγου προστασία των ζώων. Πιστεύω ότι οι κοινότητες αυτοθόνων ιδανικά θα έπρεπε να Μάλλον δεν μπορούμε να του υποχρεώσουμε να σέβονται του δικού μα κανόνε για την προστασία των ζώων. Οπότε φαίνεται να είναι απαραίτητη η απαγόρευση που έχουμε προβλέψει. Τώρα για την προστασία των ε, φυσικών θαλάσσιων πόρων, εδώ θα είμαι πολύ σαφή. Γιατί τα ζώα αυτά που έχουν θανατωθεί να ε, γίνονται αντικείμενο εμπορία. Είναι νομίζω υπερβολικό να θέλουμε να πλουτίσουμε ει βάρο του. Ξέρουμε ότι ο μόνος γνώμονας εδώ είναι το εμπορικό κέρδος. Όταν μιλάμε για χρήμα ξεχνάμε όλες μας τις αξίες και όλες μας, όλα μας τα πρότυπα. Οπότε, Πρόεδρε, συμφωνώ με την, εξε... με την κατάργηση του άρθρου 5 από τον κανονισμό, αλλά υπάρχει και η προθεσμία της 15ης Οκτωβρίου από την άλλη. Καλό θα ήταν να διορθωθεί ο κανονισμός ώστε να μην αναφέρεται ούτε έλαιο ούτε γούνα φώκες στην αγορά μας και να μην υπάρχει τέτοια δυνατότητα πριν τις 15 Οκτωβρίου. Θα πρέπει να δράσουμε άμεσα λοιπόν για να προλάβουμε στις 15 Οκτωβρίου και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε η τεχνική προσαρμογή που απαιτείται να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε οι ευρωπαϊκές αξίες και η κοινή μας ηθική να διαφυλαχθούν και να μην υπάρχουν προϊόντα από φώκια, είτε δερμάτινα, είτε γούνα, είτε έλαιο στην ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστώ κύριε Ριμπέιρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι σκότης εισηγήτρια του ΕΛΚ για την έκθεση αυτή. Και εδώ υπάρχουν τα εξή θέματα που θέλω να θέσω. Ω προ τη θέση του εισηγητή και δεδομένων των τροπολογιών 2, 3 και 5, νομίζω ότι θα πρέπει να απαγορευτεί η εισαγωγή προϊόντων φώκια που ε, παραβιάζουν τους διατάξεις του κανονισμού 2009 αλλά όχι για οποιαδήποτε χώρα εξαρτάται από τις παραβιάσεις και όχι από το από τη χώρα. Ως προς τον κανονισμό αυτών καθεαυτών έχω δύο απορίες. Ε, συγκεκριμένα στο εδάφιο 2 του τρίτου άρθρου, όπου λέγεται ότι οι περιστασιακές εισαγωγές και για κάποιο πρόσωπο μεταξύ ομάδας ταξιδοτιών ή μέλος της οικογένειάς τους. Ε, τι εννοούμε εδώ όταν υπάρχουν εμπορικοί σκοποί. Και μετά πάλι για το B του άρθρου 1, όταν μιλάμε για κοινότητες αυτοχθόνων. Δεν πρέπει να ε, οριστεί το τι εννοούμε επιβίωση και καθημερινή επιβίωση για να μπορεί να διαχωριστεί αυτό εύκολα από τους εμπορικούς σκοπούς. Δηλαδή η διατροφή και επιβίωση αυτών των κοινοτήτων. Ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ κάποια γενικά σχόλια για το θέμα της, του εμπορίου με τη, των προϊόντων φώκιας. Φυσικά ε, χαιρόμαστε για την γνωμοδότηση της, ε, της, του ΠΟΕ που επιτείνει τη δική μας απαγόρευση. Προφανώς θέλουμε να συνεχίσουμε την προστασία των ζώων. Η πρόταση της Κομισιόν η οποία τονίζει κάποιες εξαιρέσεις, ε, ε, είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και οι εξαιρέσεις για τα κριτήρια προστασίας των ζώων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρέσεις που είναι πραγματικά σημαντικές. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν και τα εισαγόμενα προϊόντα, δεν θα πρέπει να προέρχονται από εμπορικό κυνήγι, αλλά από κυνήγι για λόγους επιβίωσης. Έχουμε λοιπόν μεγάλο συμφέρον να συνεχίσουμε επικοδομητικά για την βελτίωση της πρότασης Κομισιόν και έχουμε και κάποιους ε, ορισμούς ε, για το, για το θέμα της επιβίωσης ας πούμε και για το θέμα του μη εμπορικού κυνηγιού. Αυτό νομίζω ότι θα εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις εξαιρέσεις που προβλέπονται θα μπορέσει να τη στηρίσει, τη διατήρηση δηλαδή του τρόπου ζωής ε, των αυτοχθόνων κοινωνιών και δεν θα αποτελέσει ένα βατήρα για την ε, μεταπίδηση σε ένα απλό εμπορικό ε, κυνήγι αυτού του συγκεκριμένου είδους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Ροπέ. Ε, ačiū. <clears throat> Visiškai pritariu kalbėjusiems apie draudimus, tačiau mano nuomonė. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τους ε, συναδέλφους που μίλησαν για την απαγόρευση. Από την άλλη, θα πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει παραδοσιακή μέθοδος κυνηγιού πριν ε, επιβάλλουμε απαγόρευση. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες γι' αυτό. Και επίσης πρέπει να σκεφτούμε και τις ημερομηνίες. Πότε δηλαδή θα σταματήσουν να υφίστανται αυτέ οι ε, απαγορεύσει, έτσι ώστε να έχουν απαιτούμενο χρόνο οι κοινότητε να ε, προσαρμοστούν πριν αυτή την ε, προθεσμία. Θα ήθελα να σα δώσω ένα παράδειγμα. Η Λιθουανία προστατεύει τις γκριζε φώκες γιατί πραγματικά βρίσκονται στην νομοθεσία μας, αναφέρονται ρητά και Κάθε φορά ε, βάζουμε και νέα νεογέννητες φώκες, ε, στην, ε, αφήνουμε μάλλον στο ελεύθερη στη θάλασσα. πολλές φορές έχουμε βρει στην ακτή πληγωμένες, τραυματισμένες φώκες. ερώτημα λοιπόν, οι άλλες χώρες βρίσκουν τέτοιες τραυματισμένες, πληγωμένες φώκες στις, στα παραλιά τους. Μήπως αυτό είναι αποτέλεσμα των πρακτικών κυνηγιού ή οφείλεται σε κάτι άλλο. Και σε ό,τι αφορά το 20% των εναπομεινασών φωκιών στη θάλασσα. Γενικώ εμείς είμαστε υπέρ φυσικά του να προστατεύονται οι φώκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από τις παρεμβάσεις κατανοεί κανείς ότι το θέμα αυτό του εμπορίου με προϊόντα φώκιας ουσιαστικά ε, έχει να κάνει με το πώς κυνηγούμε φώκες. Ε, είναι πάντα αρκετά ε, αντικρουόμενες οι απόψεις για το θέμα αυτό και αρκετά θερμά τα σχόλια. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του, παρόλο που δεν είναι παρόν σήμερα εδώ στην συνεδρίασή μας. Και δύο τροπολογίες θα ήθελα εγώ να υποβάλω από τη δική μας την ομάδα. Καταρχάς η έκθεση είναι πολύ καλή, πρέπει να το πω αυτό ζητά ότι μια, μια τρίτη χώρα αν δεν έχει συγκεκριμένες συμμορφούμενες αν δεν έχει προϊόντα που, που, τα κυνηγούν, που παράγονται από κυνήγι φώκιας από Ινουίτες, να μην μπορεί να τα εισάγει στην Ένωση. Αυτό καλό θα ήταν ίσως να το προτιμήσουμε αντί να έχουμε ένα εθνικό εμπάργκο. Και το δεύτερο, σε σχέση με το άρθρο 1 όπου είμαστε της άποψης ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει κατανόηση για την, παρα... για την ε, ενημέρωση ε, προς το κοινό, ενημέρωση δηλαδή των κρατών μελών για των αρμοδίων αρχών σε ό,τι αφορά τα προϊόντα αυτά, ακόμη και των τελωνιακών υπαλλήλων. Εγώ είμαι της άποψης ότι Έχουμε μια καλή πρόταση από την πλευρά της Κομισιόν, παρόλο που έχει φτάσει αρκετά αργά. Ε, είμαστε σε χρονική ε, πίεση που ε, θα, θέλαμε να μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 θα αρχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα αυτό. Και καλό θα ήταν να αλλάξουμε μόνο τα κομμάτια που έχουν τύχει επικριτικών σχολείων και από τον ε, ΠΟΕ, όχι όλο το, το σύνολο του κειμένου. Οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις συζητήσεις τις επόμενες ε, ημέρες, έτσι ώστε να έχουμε συμμορφούμενες και με τον ΠΟΕ διατάξεις και βεβαίως δεν χρειάζεται να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση για όλο το πακέτο από την αρχή. Ευχαριστώ. Ακούσαμε όλους τους βουλευτές που ήθελαν να μιλήσουν. Δεν ξέρω αν ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήθελε το λόγο επίσης. Παρακαλώ. Είστε ο διευθυντής εσείς, έτσι. Στήλστρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεσή του. Θα ήθελα να αποφεληθώ για να πω ένα-δύο πράγματα για την πρόταση που έχουμε υποβάλει. Είναι πολύ συγκεκριμένη η πρόταση. Έτσι όπως την αποστήλαμε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, με βασικό σκοπό να καλύψει τις αποφάσεις του ΠΟΕ σε συνδυασμό με το καθεστώς που ισχύει για τα προϊόντα φώκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το κάνουμε ούτως ή άλλως επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα χρειάζεται να προσαρμόσουμε την νομοθεσία μας ε, λόγω κάποιες απόφασης που προέκυψε από τον ΠΟΕ. Και χρειάζεται μια τρόπον την χειρουργική παρέμβαση για να μπορούμε να είμαστε σε ε, πλήρη συμφωνία και με τα όσα προβλέπουν οι αποφάσεις του ΠΟΕ. Εδώ προβλέπουμε τα απολύτω αναγκαία λοιπόν, ώστε να ε, ε, συνάδει πάλι η νομοθεσία μας με αυτές τις αποφάσεις του ΠΟΕ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από την σκοπιά του ΠΟΕ, έχουμε μια πολύ μακρά περίοδο για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση. Για τη δική μας βέβαια την ε, αντίληψη είναι πολύ σύντομη προθεσμία αυτή διότι μπλέκεται η διαδικασία συναπόφαση μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Θα πρέπει να έχουμε φτάσει να συμμορφωνόμαστε με την απόφαση. Όπω ξέρετε, η απαγόρευση πρώτων φώκια έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Ήδη το υπενεχθήκατε πολύ από εσά τι παρεμβάσει σα. Και η απαγόρευση αυτή που άρχισε να ισχύει το 2009 προσβλήθηκε από τον Καναδά και την Ορβηγία ε, στον ΠΟΕ ο ΠΟΕ θεώρησε ότι η απαγόρευση αυτή καθεαυτή αιτιολογείται λόγω ε, του ενδιαφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών για την καλή υγεία των φωκών. Όμως ε, ο ΠΟΕ έχει πρόβλημα με, την, ε, με τις δύο εξαιρέσεις, την εξαίρεση MRM και την εξαίρεση των Ινουιτών, σε διαφορετικό βαθμό για την καθεμία. Σε ό,τι αφορά το MRM, την κοινότητα αυτή, βρήκε οπότε ότι εδώ υπάρχει ένα εμπορικό ε, σκέλος. Δηλαδή ότι είναι διαφορετικό αυτό το κυνήγι, το κυνήγι των σκημών ε, σε σχέση με τους Καναδούς και τους Νορβηγούς. Δεν γίνεται αποδεκτή λοιπόν αυτή η απόφαση και θεωρεί ε, ότι θα πρέπει με το καθεστώς που ισχύει σε εμάς τώρα αυτό να καλύπτεται. Ο μόνος λοιπόν τρόπος να συμμορφωθούμε με αυτό το πόρισμα είναι αυτή η απαγόρευση να εξαλειφθεί από την νομοθεσία μας. Αυτό προτείναμε. Και στη φάση αυτή, επειδή το έθεσαν αρκετοί βουλευτές και σε αυτήν και σε άλλες επιτροπές αλλά και στο Συμβούλιο, ακούστηκε ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο η εξαίρεση αυτή πρέπει να διατηρηθεί. Σας διαβεβαιώνουμε ότι το εξετάσαμε από κάθε δυνατή σκοπιά και δεν νομίζουμε ότι είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Με τρόπο που να είναι νομικός ορθός. Έπειτα το πόρισμα του ΠΟΕ για την εξαίρεση των Ινουητών είναι κάπως διαφορετικό δέχεται τη διάκριση μεταξύ εμπορικού κυνηγιού, εμπορική θύρα και της θύρα των εννοητών ΟΠΟΕ λόγω των ε, κοινωνικών ε, και ιδιαίτερων συμφερόντων των Ινουητών. Εδώ το επενηθήκατε και εσείς στην σημερινή συζήτηση πριν από λίγα λεπτά, όμως Ο ΠΟΕ λέει ότι παρόλο που η εξαίρεση για τους Ινουίτες είναι αποδεκτή, ο τρόπος που έχει διατυπωθεί και οργανωθεί δεν είναι αποδεκτή. Είναι πρόβλημα ε, η ασαφής μνήμα που υπάρχει για την ε, επιμερία, την καλή για των ζώων στις ιδεολογικές σκέψεις και υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η εξαίρεση να τύχει παραβιάσεων και καταχρήσεων Η απόφαση του ΠΟΕ μα άφησε ένα μικρό περιθώριο ελιγμών για να διατηρήσουμε την εξαίρεση που θεωρούμε νίκη, νίκη για την οποία χρειάστηκε να αγωνιστούμε σκληρά. Το εκμεταλλευθήκαμε, το αξιοποιήσαμε στις συζητήσεις μας των ΠΟΕ και προτείναμε τη διατήρηση αυτής της εξαίρεσης με τρόπο ώστε όλοι οι Ινουίτες να μπορούν να την εκμεταλλευτούν. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι οι προσαρμογές αυτές έγιναν για να καλύψουμε μόνο και μόνο όσα στον ΠΟΕ, αλλά η εξαίρεση των ε, παραμένει χωρίς να πλήττεται η ε, ευημερία τους και η επιβίωσή τους και η καθημερινή τους διατροφή. Οπότε διατηρήσαμε τουλάχιστον μια εξαίρεση που έχει νόημα για τους Ινουίτες οι οποίοι έχουν αξιοποιήσει ως τώρα την εξαίρεση και θέλουμε να συνεχίσουν. Αυτά από την πλευρά μου και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς το λόγο, ο αντικαταστάτης του κ. και ο κ. Κούσμιουκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα πολύ θερμά σχόλια που εξέφρασαν για το συντάκτη της γνωμοδότησης, τον κύριο Βοητσεχόφσκι. Δεν πρόκειται να αντλήσω εγώ συμπεράσματα, πάντως σας υπόσχομαι ότι θα μεταφέρω πιστά στο συντάκτη της γνωμοδότησης όλα τα σχόλια της παρατηρήσεις και της προτάσεις σας. Ωραία. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μέχρι την 7η Μαΐου στις 12 το μεσημέρι προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, ολοκληρώνω αυτό το σημείο. Έχετε λάβει με mail αλλά και ε, εγγράφος της ε, αποφάσης των συντονιστών και τις σχετικές πληροφορίες από την συνεδρία των συντονισμών των συντονιστών, συγγνώμη. Έχετε λοιπόν τις συστάσεις τις προτάσεις και τις αποφάσεις των συντονιστών και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις θεωρώ ότι τις εγκρίνουμε. Διεκπαιρεώσαμε το πρόγραμμα εργασιών μας, πλησιάζουμε προς το τέλος της συνεδρίασης μετά από μια μισή ώρα απογευματινής συνεδρίας καταφέραμε σε μια μισή ώρα να διεκπαιρεώσουμε όλα τα απογευματινά μας θέματα. Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι καλό απόγευμα. Ραντεβού στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής της 26 Μαΐου που θα γίνει παρουσία και του Επιτρόπου Χόγκαν. Οπότε αν έχετε ρωτήσει παρατηρήσεις ε, σκεφτείτε τα και στείλτε τα από τις πολιτικές ομάδες στη Γραμματεία για να τις διαβιβάσουμε στον ε, Επίτροπο ώστε να είναι προετοιμασμένος ε, για το διαρθρωμένο διάλογο και να μπορέσουμε με τις ερωτήσεις μας να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Σας ευχαριστώ θερμά. Ραντεβού στην επόμενη συνεδρίαση. Χαίρετε.